Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ε, κοινοποιήσω ορισμένες ε, προφορίες. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ελπίδα μου ότι η συνεργασία μου με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας θα καρποφορήσει. Διότι ξέρετε ότι σε μία εβδομάδα τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη Λισαβόνας. Ελπίζω όλα αυτά να προχωρήσουν απρόσκοπτα. Ε, σε σχέση λοιπόν με το θέμα αυτό. Είμαι σε μόνιμη επαφή με το πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τους εκπροσώπους της ε, Σουηδικής ε, Προεδρίας. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρόθυμο να κάνει τις ακροάσεις των υποψηφίων ε, επιτρόπων και έχω ενημερώσει και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο και ε, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άλλο θέμα. Την άλλη εβδομάδα, την 1η ε, Δεκεμβρίου, γνωρίζετε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνετε το κοινό για το AIDS για να αυξάνεται και τα πολέμηση. Στη συνέχεια, Έχουμε την 65η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ομόφωνα έγινε δεκτή αυτή η διακήρυξη και ήταν πραγματικά το πρώτο σημαντικό επίτευγμα ε, του ΟΗΕ ε, στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να σας πω ότι για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η επέτειος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα ο μέλημά μας. Ε, προχωρώ τώρα στα συνοπτικά πρακτικά ε, που διανεμήθηκαν τις 12 Νοεμβρίου και τα κείμενα που εγκρίθηκαν τότε. Έχετε λάβει τα συνοπτικά πρακτικά, δεν ξέρω